liebe Kollegen und Ο Πρόεδρος, ας αρχίσουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Τώρα, για την ημερησία διάταξη. Έχετε τροποποιήσεις να προτείνετε. Όχι. Καλά λοιπόν. Τότε. Η ακρόαση που είχε προβλεφθεί για αύριο αντίκτυπο ειδική ομάδα τη Επιτροπή όσον αφορά την διαδικασία μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα μετά από απέτηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά από συζήτηση με τους Προέδρους των πολιτικών ομάδων, μετά από προβληματισμό που προέκυψε χθες και για λόγους αρμοδιοτήτων, αναβλήθηκε. Έχω ενημερώσει τους συντονιστές. Προσωπικά δηλώνω ότι σχετικά με τα επιχειρήματα του Προέδρου Έχω βεβαίω κατανόηση ότι ωστόσο η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού θεωρεί παρά ότι το θέμα της αντιμετώπισης των δαπανών στην Ελλάδα και γενικά της διαχείρισης των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα αυτή σαφώς εμπίπτουν σύμφωνα με το άρθρο 7 στο πεδίο αρμοδιότητας της παρούσας Επιτροπής και γι' αυτό στην συνεδρία των συντονιστών αποφασίσαμε να αναβάλουμε την ακρόαση, αλλά το δυνατόν συντομότερο θα διεξαγάγουμε τη συζήτηση αυτή με εκπροσώπους της Task Force και θα προετοιμαστεί δεόντως. Τώρα, η παρούσα συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Κάθε ένας λοιπόν από εσά που λαμβάνει το λόγο και πατά το κουμπί του μικροφόνου μπορεί ε, να, μπορούν να τον βλέπουν σε ολόκληρο το διαδίκτυο. Τότε, θα έρθω λοιπόν στην ημερήσια διάταξη και δει στο υπαριθμό τέσσερα θέμα της ημερησία διατάξεως που αναφέρεται στη χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινή γεωργική πολιτικής. Η εισηγήτρια είναι η κυρία Ηλιάνα Ιβάνοβα. Α, μια στιγμή διορθώνω, έχει αναβληθεί διότι η κυρία Ιβάνοβα είναι απούσα. Δώστε μου παρακαλώ την επικαιροποιημένη ε, ημερησία διάταξη. Αρχίζουμε λοιπόν με το θέμα υπαριθμών 6. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής στον πυρηνικό σταθμό της Ιγναλίνα στην Λιθουανία. Έχετε το πρόγραμμα μπροστά σας. Θα μπορέσουμε να διεξαγάγουμε λοιπόν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις Επ' αυτών των θεμάτων υπάρχει κανείς που επιθυμεί να λάβει το λόγο. Όχι. Καλά λοιπόν. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίνεται το πρόγραμμα της επισκέψεως αυτής και επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε σε άλλο θέμα της ε, ημερησίας διατάξεως. Äh, ist Είναι δυνατόν βέβαια ο κ. εκπρόσωπο εκπρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου, να λάβει το λόγο και να μα εξηγήσει. Κύριε Φαζάκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ε, ευγενή σας καλοσύνη να με προσκαλέσετε. Μπορώ να σας δώσω ορισμένες, αν θέλετε, συμβουλές ή υποδείξεις για την ε, επίσκεψή σας στην Λιθουανία. Επιτρέψτε μου πρώτα να σας δώσω μια σύνοψη της καταστάσεως και να τονίσω ορισμένα πράγματα που νομίζω ότι θα έπρεπε να βάλετε στις αποσκευές σας για την αντιπροσωπή αυτή. Πρώτα λοιπόν κυρίες και κύριοι αγαπητά μέλη θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού που με προσεκάλεσε στη σημερινή ανταλλαγή απόψεων για την προπαρασκευή τη ε, μετάβαση αντιπροσωπεία στον πυρηνικό σταθμό τη Ιγναλίνα στην Λιθουανία. Είναι ορθή η ε, προσέγγιση σας στα θέματα αυτά και η απόφασή σας επίσης να μεταβείτε στην Λιθουανία που βέβαια έχει σχέση με το πρόγραμμα αφοπλισμού των πυρηνικών σταθμών. και δίνεται και κοινοτική ενίσχυση στην Λιθουανία και στη Σλοβακία από την Ένωση για τον παροπλισμό μάλλον των πυρηνικών εργοστασίων. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να κλείσουν τα εργοστάσια αυτά νωρίτερα. Τώρα, το ίδιο το πρόγραμμα παροπλισμού, το βασικό μας συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει ήδη ένα πρόγραμμα βασισμένο στις ε, σχετικές μελέτες και η απόφαση για το μέγεθος και τον χρονισμό των μελλοντικών χρηματοδοτήσεων στο λείπει. Ο βασικός στόχος της αρχικής μας ε, μελέτης, έρευνας δηλαδή, ήταν το ίδιο το decommissioning, ο παροπλισμός και επισκεφθήκαμε τις χώρες για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Η Λιθουανία ήταν πρώτη και πιο σημαντική χώρα και επομένως στο σχεδιασμό της επίσκεψη αντιπροσωπεία σα, μπορείτε να βασιστείτε στην εκθεσή μα, η οποία θα σα δώσει και το ιστορικό και την ανάλυση των γενικών τάσεων και γεγονότα, καθώ επίση και τα όσα έχουμε συλλέξει από την έρευνά μα. Δύο χρόνια λοιπόν μετά από την έρευνα, αυτόν τον έλεγχο που διεξάγαμε εκεί, μπορείτε να ελέγξετε τι τάσει αυτέ και κατά πόσον ε, εφαρμόστηκαν οι συστάσεις. Και εσείς που είστε το πολιτικό όργανο που δίνει την έγκριση μπορείτε να συναγάγετε τα συμπεράσματά σας για τις μελλοντικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Τώρα, λεπτομέρειες για το πρόγραμμα παροπλισμού και την εφαρμογή στη Λιθουανία. Η έκβαση του προγράμματος παροπλισμού μετά από την δαπάνηση 1,3 δισεκατομμυρίων ε, ευρώ δεν έχει επιτύχει τους στόχους του. Έχουμε ακούσει και φωνές πρόσφατα για την επανέναρξη ε, ε, λειτουργίας. Εντοπισμός των δραστηριοτήτων και των τεχνολογιών πρέπει να γίνει ακόμη. Βασίζεται ε, στις στρατηγικές και στον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων το, ο προγραμματισμός στην χώρα αυτή είναι πολύ περίπλοκος και έχει πολλές πτυχές και επίπεδα. Αλλά δεν υπάρχει επαρκής παρακολούθηση. εξαρτώνται ακόμα από εξωτερικούς συμβούλους. Αυτό που χρειάζεται περισσότερη εξήγηση, για όλους μας δηλαδή, είναι να δημιουργηθεί το management δύο διάβλων, που είναι η δίκευση της ε, Λιθουανίας. Έχει οδηγήσει όμως σε επικαλύψεις, έλλειψη πληροφοριών, ε, ανευθυνότητα, καθυστερήσεις ε, στον παραπλησμό και έλλειψη διαφάνειας. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί τι, ποιος ήταν και ποιος θα είναι ο ρόλος της τράπεζας αποκατάστασης, μάλλον στη Λιθουανία. Προτάσεις σχετικά με το μέλλον του προγράμματος ε, παροπλισμού βασίζονται στην έκθεσή μας και στην πρόταση της Κομισιόν που προβλέπει η Λιθουανία να υποβάλει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα παροπλισμού μέχρι το 2014. Θα πρέπει να θεσπιστούν οι ευθύνε και μεταξύ 2014 και 2017 προβλέπονται 219 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυση προς τη Λιθουανία για τον παροπλισμό της Ιγναλίνα. Αντιθέτως τώρα το Υπουργείο Ενέργειας της Λιθουανίας θεωρεί ότι οι ανάγκες χρηματοδοτήσεως των δραστηριοτήτων παροπλισμού για τα έτη 2014 έως 20 ανέρχονται σε 870 εκατομμύρια ευρώ και γι' αυτό ζητούν 770 εκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για το πρόγραμμα αυτό. Είμαι πεπισμένος ότι η επικείμενη επίσκεψή σας θα παίξει σημαντικό ρόλο. Εάν θεωρήσετε αναγκαίο να εξετάσετε ορισμένες πτυχές του προγράμματος στα πλαίσια της συνέχειας της ε, εξέτασής μας, του ελέγχου μας, ασφαλώς και θα συνεργαστούμε με το ευρύτερο δυνατό πνεύμα. Σας εύχομαι καλή επίσκεψη, το έγγραφό μας είναι στη διάθεσή σας και αναμένουμε με ενδιαφέρον και ανυπομονησία να συνεργαστούμε μεταξύ σας. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας υποβάλω τις προτάσεις αυτές. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Φαζάκας. Και εξ ονόματος ε, της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολισμού ευχαριστώ το ελεγκτικό συνέδριο. Οι εκθέσεις του είναι πολύτιμες και έχει μεγάλη σημασία τώρα βέβαια που τους δώσατε επίκαιρη μορφή. Δεν είναι εύκολο το θέμα αυτό. Πριν θέσω υποσυζήτηση την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου θα ήθελα να παρακαλέσω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ή μάλλον την εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ή μάλλον όχι τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, αν θέλει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τον προγραμματισμό της επισκέψεώς σας. Επιτρέψτε μου πρώτα μία γενική παρατήρηση με το πρόγραμμα της επισκέψεως θα καλύψετε το πυρηνικό, την πυρηνική πτυχή, τα προγράμματα ενέργειας τα οποία έχουν ήδη κινηθεί για, έχουν ήδη ξεκινήσει για να αντισταθμίσουν το κλείσιμο, δηλαδή ε, εγκαταστάσεις αποθειώσεως και καύσος αερίου κλπ. Αυτά δεν θα τα δείτε Επομένως, δεν θα δείτε πού πηγαίνουν περίπου 30% των χρηματοδοτήσεων. Για την εγκατάσταση Γναλίνα την ίδια, εμείς στην πρώτη έκτου κάναμε διάσκεψη δωρητών στο Λονδίνο, η οποία διάσκεψη δωρητών αναγκάστηκε να διαπιστώσει με λύπη της ότι για ένα έργο κλειδί δεν μπορεί να σημειώσει επαρκή πρόοδο, ικανοποιητική πρόοδο. Και το έργο Β1, Interim Fuel Storage Facility, παίζει ε, ρόλο κλειδί διότι το έργο αυτό οφείλει να υλοποιηθεί έτσι ώστε να μπορέσει να κενωθεί από το σχάσιμο υλικό ο δεύτερος Πυρηνικό αντιδραστήρα. Ο πρώτο είναι η διάδιος, Οι δραστηριότητε παροπλισμού γίνονται, λαμβάνουν χώρα γύρω από τον αντιδραστήρα αυτό. Ο δεύτερος αντιδραστήρας, όπως και η δεξαμενή ψήξεω, είναι ακόμη πλήρη, είναι γεμάτε. Και γι' αυτό πρέπει να δημιουργηθεί η κατάσταση προσωρινής αποθήκευση ε, του σχάσιμου υλικού και μόνο όταν ο δεύτερο αντιδραστήρα θα είναι κενός, μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτά που είπε ο κύριος Φαζάκας, δηλαδή μη αναστρεψιμότητα της διαδικασίας. Ως γενική πληροφορία ήθελα να σας θέσω υπόψη να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή όταν θα είστε επί σε αυτό το ε, συμπληρωματικό έργο το οποίο βέβαια παίζει κέριο ρόλο για το σωστό χρονισμό της όλης προσπάθειας. Ευχαριστώ για τη σημαντική αυτή πληροφορία. Υπάρχουν παρατηρήσεις ή σχόλια από την Επιτροπή. Ο κ. Γκάιερ. Εάν εξετάσουμε τη συνολική εικόνα σχετικά με τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου στις διαπραγματεύσεις για το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο με τις χώρες μέλη ασχολούμεθα τώρα να βρούμε πόσα μπορεί να δαπανά η Ένωση από το 2014 και μετά. Η ερώτησή μου προς εσάς τους δύο που μιλήσατε πριν είναι εν ώψη του ιστορικού παραμένω στο παράδειγμα του σταθμού Ιγναλίνα σε ό,τι αφορά το ύψος της των δαπανών αυτών, μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το ύψος του ποσού το οποίο ενδεχομένω θα χρειαστεί να δαπανηθεί ακόμη έτσι ώστε να παροπληστεί τελεσίδικα ο σταθμός αυτός και κατά πόσο αποτελεί κίνδυνο για τον προπολογισμό με την έννοια ότι ίσως να προκληθούν να προκληθεί μεγαλύτερο κόστος έτσι ώστε από το 2014 και μετά να ε, ε, έχει συνέπειες για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρόεδρος, άλλες ερωτήσεις ή τοποθετήσεις. Από ό,τι βλέπω όχι. Κύριε Φαζάκας. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όπως επιβεβαιώθηκε και στην εκθεσή μας, όπως άλλωστε περιλαμβάνεται και στην γνωμοδότηση της Κομισιόν για την έκθεσή μας, θα πρέπει η Λιθουανία να υποβάλει ένα ξεκάθαρο λεπτομερές σχέδιο για τον παροπλισμό, το χρονικό επιμερισμό καθώς και το κόστος. Αυτά θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι το 2014. Για την ώρα έχουμε μοναχά ένα σχέδιο της Λιθουανίας, το οποίο σχέδιο προβλέπει από ότι από το 2014 έως 20 ολόκληρο αυτό το έργο, το σχέδιο, θα ανέλθει περίπου στα 900 εκατομμύρια ευρώ. Ακριβέστερα 870 εκατομμύρια ευρώ. Και από αυτά τα χρήματα η Λιθουανία απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυση 770 εκατομμυρίων ευρώ. Για την περίοδο αυτή όμως η Κομισιόν προβλέπει μόνο 229 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό χρηματοδοτικό κενό και λέμε ότι η απόσταση από τα διαθέσιμα μέχρι τα ετούμενα ποσά είναι σημαντική. Γι' αυτό, όπως ρωτήσατε και εσείς, πρέπει να ρωτήσετε πότε θα υπάρχει πλήρης τελικός σχεδιασμός πρέπει να αναφερθούν συγκεκριμένα ποσά και μετά βέβαια θα είναι απαραίτητο να γίνει ένα σκληρό γύρος διαπραγματεύσεων Ποιο θα χρηματοδοτήσει τα ποσά αυτά. Καταρχήν εμείς ε, θεωρούμε ότι ισχύει η αρχή του ορυπαίνων πληρώνει. Αυτοί θα πρέπει να πληρώσουν λοιπόν. Όμως, όπως με επιτρέψατε να σας πω και προηγουμένω. Πρόσφατα ακούσαμε από Λιθουανούς πολιτικούς και άλλες προσωπικότητες ότι εάν η χρηματοδότηση δεν είναι επαρκής, σκέπτονται, λένε, να ξανανοίξουν τον πυρηνικό σταθμό. Ενώ η Κομισιόν μιλάει για μη αντιστρέψιμο τη διαδικασία παροπλισμού. Άρα θα πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή σε ένα σημείο όπου η χρηματοδότηση να μην διασυνδέεται με τον κίνδυνο να ανακοπεί η πορεία του σχεδίου παροπλισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να συζητηθεί τόπου με τις αρμόδιες λιθωνικές αρχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φαζάκας. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Άλλος κανείς δεν μου έχει ζητήσει το λόγο. Και άρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και προχωρούμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως και αφού είναι ακόμη απούσα η κυρία Ιβάνοβα, προτείνω να έλθουμε στην γνωμοδότηση του κυρίου Ντόιτς, να συμφωνεί ο συναδελφός μας λοιπόν, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί καλεσμένοι και ακροατές. Το σχέδιο γνωμοδότησή μου αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το σχετικό κανονισμό, τη σχετική πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ενισχύσεις αυτές. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία σημεία της γνωμοδότησης. Καταρχήν να σας κάνω μια γενική ανασκόπηση αυτού του σχεδίου της πρότασης κανονισμού. Να σας περιγράψω λίγο το ιστορικό υπόβαθρο και να αναφερθώ και σε δύο άλλα σημεία. Η προτάσει για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής εκπονήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Γεωργίας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταρτίζει έκθεση ως αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή. Η δική μας Επιτροπή, η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού, καλείται να γνωμοδοτήσει στην ε, έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας. Η Επιτροπή Γεωργίας, λοιπόν, με εισηγητή τον κύριο Λαβία, εκπονεί σχετική έκθεση και μάλιστα και το ελεγκτικό συνέδριο θα δώσει τη δική του γνωμοδότηση. Εμείς στην Επιτροπή μας διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό σφαλμάτων στις ενισχύσεις για τη γεωργία δεν είναι υπερβολικά υψηλό. Και οι τελευταίες τρεις εκθέσεις ε, του ελεκτικού συνεδρίου δίνουν ε, ένα συντελεστή σφάλματος 2,3%. Δηλαδή πολύ κοντά στο στόχο που είναι το 2% ποσοστό σφάλματος. Σε ό,τι αφορά τις βασικές προτάσεις της γνωμοδότησής μου, όπως είπε και ο κύριος ε, Κρετά, στην τελευταία συζήτηση που είχαμε επί της εκθέσεως του ελεκτικού συνεδρίου. Έχουμε τρία κυρίως σημεία, γύρω από τα οποία περιστρέφεται και η δική μου γνωμοδότηση. Καταρχήν, ποιοι είναι οι στόχοι που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για τον κανονισμό αυτό. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να είναι ε, πιο συγκεκριμένη και οι έλεγχοι και οι να είναι πιο διαφανείς και πιο αποτελεσματικοί. Επίσης, υπάρχει και το θέμα της απλούστευσης που είναι ζητούμενο στην πρόταση κανονισμού. Δεν θα ήθελα να επισέλθω στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης μου γιατί έχετε λάβει και το κείμενο, οπότε δεν έχει νόημα να μακρηγορώ. Θα ήθελα πάντως να πω ότι συμφωνώ με τις ε, δηλώσεις και τα συμπεράσματα του ελεκτικού συνεδρίου ως προς τους στόχους. Δηλαδή ότι οι στόχοι και οι σκοποί της πρότασης κανονισμού χρήζουν περαιτέρω ε, προσδιορισμού και συγκεκριμενοποίησης, γιατί είναι κάπως ε, αόριστη αυτή τη στιγμή. Εξού και οι τροπολογίες που κατέθεσα και που έχουν στόχο να διευκρινίσουν τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να καταστήσουν πιο συγκεκριμένους αυτούς τους στόχους του κανονισμού, πιο αποτελεσματικούς και πιο σαφείς. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις, και εδώ είναι σημαντικό να είναι υποχρεωτική. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη θα πρέπει στα προγράμματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου να υπόκειται σε έλεγχο ως προς την εφαρμογή. Και θα πρέπει πριν την έγκριση των προγραμμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, βεβαιώνεται ότι τα κράτη-μέλη έχουν σαφείς μηχανισμούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επαλήθευσης και ελέγχου ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος αυτών των προγραμμάτων και να περιορίσετε το ποσοστό σφαλμάτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απλούστευση, είμαι και εγώ υπέρ της απλούστευσης, αλλά θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε ως σύνθημα. Γιατί είναι αξιέπαινος ο στόχος της απλούστευσης, αλλά δεδομένου ότι έχουμε μία επταετία μπροστά μας ως προς το πλαίσιο, θα πρέπει η απλούστευση αυτή να έχει μία αντανάκλαση και στις διατάξεις και στους εφαρμοστικούς κανόνες. Οι τροπολογίες 7 και 13 στόχο έχουν την ε, ενίσχυση αυτής της απλούστευσης ώστε να ωφελούνται και οι τελικοί χρήστες του κανονισμού. Προτείνουμε και μια μεγαλύτερη διαφάνεια των διοικητικών διατυπώσεων που προτείνουμε να γίνουν και πιο φιλικές προς το χρήστη. Έχω καταθέσει και τρεις τροπολογίες πιο τεχνικού χαρακτήρα με βάση τα πορίσματα του ελεγκτικού συνεδρίου και αυτό που μας είπε ο κύριος Κρετά στην προηγούμενη μας συνάντηση θα πρέπει να γίνουν πιο διαφανείς αποδοτικοί και αποτελεσματικοί έλεγχοι και το όλο σύστημα να γίνει πιο απλό. Αυτή είναι η ζητούμενη στόχη και από τις τροπολογίες μου. Äh, Ευχαριστώ κύριε Ντόιτς. Από την, γενική, ε, από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν έχετε το λόγο κύριε Γενική Διευθυντά. μπορείτε να πείτε την άποψή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε συντόμως. Θα είμαι όπως είπα σύντομος. Για κάθε μια από τις τροπολογίες έχουμε βέβαια ειδικότερε παρατηρήσεις, αλλά νομίζω θα ήταν υπερβολικό να μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Θα αναφερθώ στα τρία θέματα που έθιξε ο εισηγητής και θα κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Πρώτα για τους στόχους. Νομίζω ότι στην αξιολόγηση προτάσεως της Κομισιόν έχουμε σαφώς μια απόκληση απόψεων. Η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει η πολιτική αναπτύξεως της υπαίθρου να προσανατολίζεται σε έξι προτεραιότητες, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την επίτευξη ο σκοπό μάλλον την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020. Αυτές οι εξωτερότητες υποδιαιρούνται σε 18 επιμέρους στοχεύσεις που αποτελούν ένα είδος ε, κατευθυντήριων γραμμών για τις χώρες μέλη. Συνολικά πρέπει να πει κανείς ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου βασίζεται σε μια σταδιακή προσέγγιση η οποία λειτουργεί εκ των κάτω και όχι εκ των άνω. Δηλαδή δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη η οποία υπαγορεύει στις χώρες μέλη την πολιτική ανάπτυξη της Πέθρου. Οι χώρες μέλη θα ακολουθούν μια ανάλυση που λέγεται SWOT και η οποία αναλύει τις ανάγκες επιτόπου. Στη βάση αυτής της αναλύσεως θα καταγράφουν τις ανάγκες ε, των περιφερειών αλλά και των χωρών μελών. Το να προβλέψουμε εδώ ειδικότερου στόχους μέχρι και επίπεδου επιμέρους δράσεων πιστεύω ότι θα ήταν αντίθετο στην ιδέα της ε, περιφερειακής ανάπτυξης και δεν θα επέτρεπε στους χώρους, στις χώρες μέλη να επιτύχουν τους στόχους αυτούς. Γι' αυτό για τις τροπολογίες 2, 4 και 6 δηλώνουμε ότι μας προκαλούν προβλήματα. Δεν θα πω στις λεπτομέρειες τώρα, αλλά σημειώνω, όπως είπα πριν, ότι δυσκολίες μας προσκαλούν οι τροπολογίες 2 4 και 6. Συμφωνούμε κατά τα άλλα με την άποψη του εισηγητού ότι πρέπει να είναι εξασφαλισμένη μια καλή διαδικασία προγραμματισμού και επομένως και η διαχείριση αυτή πρέπει να παρακολουθείτε και να εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο προγραμματισμός, ωστόσο, στα πλαίσια της κοινή διαχείρισης των ε, δαπανών, ανατίθεται στις χώρες μέλη. Και καθήκον της Κομισιόν είναι να εξετάζει τα προγράμματα που βάλουν οι χώρες μέλη. Αυτό άλλωστε περιλαμβάνεται και στην πρόταση της Κομισιόν, όχι μόνο ως δυνατότητα, αλλά και ως καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά την εποπτεία της παρακολούθησης της εφαρμογής των προγραμμάτων, εδώ δεν κινούμεθα τόσο μέσα στα πλαίσια της πρότασης της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου, αλλά περισσότερο στα πλαίσια του λεγόμενου οριζόντιου κανονισμού, που προβλέπει τις λεπτομερέστερες διατάξεις ιδίως σχετικά με τους ελέγχους αλλά και για την εκροή των κονδυλίων εφόσον τέτοια δεν ε, έχουν δοθεί αλλά όχι σε συμφωνία με τους ε, κανόνες της Ένωσης. Έρχομαι σε ένα επιμέρους θέμα εδώ. που περιλαμβάνεται στην πέμπτη τροπολογία και αναφέρεται στην εξασφάλιση από πλευράς Κομισιών ότι έγινε σωστά η εθνική διαδικασία πιστοποίησης. Εδώ ο τομέας αυτός εντάσσεται στην πραγματικότητα στον οριζόντιο κανονισμό. Και θεωρούμε ότι στα πλαίσια της κοινή κατανομής των αρμοδιοτήτων δεν μπορεί να αποφασίζεται από την Κομισιόν, παρά μόνο η Κομισιόν μπορεί να κρίνει εκ των υστέρων αν οι αποφάσεις των χωρών μελών ήταν ορθές και να εξάγει τα αντίστοιχα συμπεράσματα. και όταν υπάρχουν και 81 οργανισμοί πληρωμής, αντιλαμβάνεστε ότι η η εποπτεία δεν είναι δυνατή. Εξάλλου η πρόταση της Κομισιόν περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία, ιδίω την, την καταποκοπή συνολική ε, υπολογαριασμών για το κόστος. Εκεί μπορεί να γίνει σημαντική απλούστευση Τέτοιε προτάσει περιλαμβάνονται στο οριζόντιο κείμενο το οποίο ισχύει για όλα τα διαρθωτικά ταμεία και έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κανονισμό για τι κοινέ διατάξει όλων των διαρθωτικών ταμείων που βέβαια δεν αποτελεί αντικείμενο τη παρούση εκθέσεω, αλλά βέβαια και αυτά τα στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και γι' αυτό νομίζουμε ότι το σχέδιο εκθέσεω αποτελεί καλή βάση για την συζήτηση αλλά βεβαίω υπάρχουν ορισμένα επιμέρου θέματα όπου θεωρούμε ότι οι προτάσεις του εισηγητού δεν ανταποκρίνονται στις προθέσεις, στις πολιτικές προθέσεις όπως αυτές έχουν περιληφθεί στην αρχική πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Βέγγελε. Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση θα ήθελα να απευθύνω το καλό ορίσατε στον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου και να τον ρωτήσω αν επιθυμεί να λάβει το λόγο. Όχι. Καλά λοιπόν, ο κύριος Ιβαν. Ο κύριος Ιβαν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Ντόιτς, γιατί έχει βελτιώσει κατά πολύ τη γνωμοδότησή του. Έχουμε κάποιες τροπολογίες, την 8 και την 9 για παράδειγμα, που αναφέρονται στους μικρούς καλλιεργητές και δεν συμφωνώ με την πρόταση διαγραφής των δύο παραγράφων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο επικοδομητικοί και να ζητήσουμε περισσότερες διευκρινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων. Σίγουρα δεν μπορούν να μείνουν αμετάβλητες οι δύο παράγραφοι, θα πρέπει να αναδιατυπωθούν, αλλά δεν συμφωνώ με τη διαγραφή τους. Δεν νομίζω ότι μία ολοσχερής διαγραφή των παραγράφων θα λύσει το πρόβλημά μας. Προτιμώ να ζητήσουμε εξηγήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για την τροπολογία 12, που αφορά την έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων αποφάσεων και επενδυτικών αποφάσεων. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε πιο μετριοπαθείς να ζητούμε μελέτη επιπτώσεων που θα ευθυγραμμίζεται με την ε, παρούσα νομοθεσία. Ένα άλλο πρόβλημα αφορά τους δικαιούχους ενισχύσεων για ιδιοκτήτες δασών. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, έχουμε πολλές ε, τοπικές ε, κοινότητες που είναι ιδιοκτήτες δασών, αλλά δεν είναι επιλέξιμοι για τέτοιες ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. γιατί μιλούμε για, τις, ε, για τους περιορισμούς που επιβάλλει το πρόγραμμα Natura 2000. Θα πρέπει και αυτά τα σημεία να τα λάβουμε υπόψη. Θα ήθελα πάντως να ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή μας και να ζητήσω να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι και οι ιδιώτες και οι δικαιούχοι δημοσίου θα κάνουν παρόμοια πράγματα. Οπότε θα πρέπει και το δημόσιο να δικαιούται και να είναι επιλέξιμο για επιδοτήσει, όπω και οι ιδιώτες. Ο εισηγητή επιθυμεί να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, κύριε και κύριοι. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ε, μοιραστήκατε μαζί μου τις απόψεις ε, και για τις επικοδομητικές σας συμβουλές. Έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Καταρχήν πιστεύω πως χρειάζονται περαιτέρω διαβουλεύσεις. ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη τα επιχειρήματα της Κομισιόν και να προσπαθήσουμε να τα εναρμονίσουμε με τις απόψεις και την γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Πιστεύω πως η επικουρικότητα μάλλον πιστεύω στην επικουρικότητα και στην ανάπτυξη από κάτω προς τα πάνω και γι' αυτό και στηρίζω την πρόταση της Κομισιόν. Από την άλλη πλευρά πιστεύω πως χρειάζεται να εστιάσουμε στο τελικό χρήστη και να έχουμε στόχους που να είναι επιλέξιμοι, αποτελεσματικοί και αποδοτικοί. είναι γνωστό ότι ε, όταν ευαισθιαζόμαστε σε λιγότερα πράγματα πετυχαίνουμε περισσότερα γι' αυτό και έχουμε έξι τομείς προτεραιότητας ε, Νο, υπάρχουν κάποιοι στόχοι που δεν είναι συμβατοί που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Κομισιόν και αν και μιλάμε για πολιτική συνοχής και για ανάπτυξη της υπαίθρου Αυτά είναι παρόμοια, αλλά φυσικά όταν κάνουμε συγκρίσεις μπορεί να κάνουμε και λάθη. Και στην ε, πολιτική συνοχή εστιαζόμαστε σε, θέματα, ε, σε θεματικούς τομείς, ενώ εδώ μιλάμε για στόχους. Οπότε δεν συνδυάζονται αυτά. Όσον αφορά τους ελέγχους, την παρακολούθηση, αληθεύει ότι οριζόντια προσέγγιση μπορεί να μας δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, ωστόσο επί τη βάση της εμπειρίας μας βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη υποβάλλουν τα προγράμματα για ανάπτυξη υπαίθρου, η Κομισιόν τα εγκρίνει και μετά όταν ε, γίνονται έλεγχοι τότε η Κομισιόν βλέπει προβλήματα στην ε, ε, διαπίστευση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρούμε μια καλύτερη λύση από την άποψη των κρατών μελών και ότι πριν να εφαρμοστούν τα προγράμματα θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια ε, διαπίστευσης. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε λιγότερο διοικητικό φόρτο και ότι το ολόκληρο το πρόγραμμα θα μπορούσε να είναι πιο ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό. Ελπίζω λοιπόν ότι τελικά θα φτιάξουμε μια πολύ καλή κοινή γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ε, τροπολογίες μέχρι τις 10 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου. Εδώ λύγει το θέμα αυτό της ημερησίας διατάξεως και ευχαριστώ όλες και όλους όσοι έλαβαν το λόγο. Ερχόμαστε στο 4 τώρα. Η κυρία Ιβάνοβα έχει προσέλθει και την καλωσορίζω και της δίνω ευθύς αμέσως τον λόγο η κυρία Ιλιάνα Ιβάνοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Μόγκελε, και τον κύριο Κρετάν από το Ελεκτικό Συνέδριο για την πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Θα ήθελα να αναφερθώ στα πιο κέρια σημεία αυτής της πρόταση κανονισμού. Καταρχήν χρειαζόμαστε σαφείς δείκτες, στόχους και ε, περισσότερες διατάξεις για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Ε, δεύτερο, το θέμα της προφύλαξης και της πρόληψης. Ε, εγώ είμαι υπέρ της πρόληψης. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προφύλαξης, γιατί το φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Είναι πολύ πιο εύκολο να προλάβουμε παρά να χρειαζόμαστε πιο δαπανηρά μέτρα. Επίσης θα πρέπει ε, οποιαδήποτε αύξηση της χρηματοδότησης ε, να αιτιολογείται δεόντως και να υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα και σε ό,τι αφορά την απλούστευση. Συμφωνώ με την απλοποίηση των διαδικασιών, αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να είμαστε απρόθυμοι σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της παρακολούθησης και του ελέγχου. Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω τα βασικότερα στοιχεία των τροπολογιών, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, ό,τι αφορά τι εξουσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε τελικό λόγο αρμόδια για την εκτέλεση του προπολογισμού και την αποτελεσματική αξιοποίηση των και εφαρμογή των δαπανών. Γι' αυτό θα πρέπει να έχει ένα αποπτικό ρόλο σε ό,τι αφορά στη διαδικασία διαπίστευση των οργανισμών πληρωμής. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ε, υπερβολικά εκτεταμένης χρήσης των καταποκοπήν διορθώσεων. Επίσης, ε, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναθεωρήσει το σύστημα ε, των οργάνων πιστοποίησης και των επιδόσεων τους, προκειμένου να γίνει αποτελεσματικό το έργο αυτών των οργανισμών πιστοποίησης. Συμφωνώ και με τα πορίσματα και τα σχόλια του ελεκτικού συνεδρίου για το θέμα αυτό. Επίση, σημαντικό θα είναι να διευκρινίσουμε ότι οι έλεγχοι τη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οργανισμού Πληρωμή και στου φορείς πιστοποίηση θα πρέπει να στηρίζονται ε, στους κινδύνους. Έτσι θα μειωθεί το διοικητικό άχθο ε, και θα κρατήσουμε ένα επαρκέ επίπεδο ελέγχου. Άλλη σημαντική κατευθυντήρια γραμμή των τροπολογιών είναι η αύξηση της ε, ενίσχυση της διαφάνειας. Οι φορείς πληρωμής θα πρέπει να έχουν σαφή κριτήρια και ε, στόχους ώστε να μπορούν να, δίνουν, να κάνουν αναφορά και να είναι υπόλογε για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίζει σαφείς, ε, σαφείς στόχους και σαφή κριτήρια. Επίσης τα, θα πρέπει να δημοσιεύονται τα πορίσματα, τα συμπεράσματα των οργανισμών πιστοποίησης και αν ε, δίνουν σαφή διαχειριστική ε, δήλωση αξιοπιστία, θα πρέπει να μπορούν να υπολογίζουν τα επίπεδα σφάλματο που δημοσιοποιούνται. Και τέλο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει σαφεί και εναρμονισμένου κανόνε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή των τόκων για τα χρέη για τα κρεμή χρέη. Σε ό,τι αφορά τι κατεξουσιοδότητε πράξη, πιστεύω ότι θα πρέπει εδώ να εξασφαλίσουμε και το ρόλο του ελεκτικού συνεδρίου με, το 200, με βάση το άρθρο 290 τη συνθήκη. Θα πρέπει η Επιτροπή να έχει αρμοδιότητες για κατεξουσιοδότηση πράξη με βάση τον οριζόντιο κανονισμό, αλλά θα πρέπει και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαμορφώνουν γνώμη με βάση τη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη του ελεκτικού συνεδρίου. Επίση, το ελεκτικό συνέδριο θα μπορούσε να προσκαλείται και να εκτιμά τα κριτήρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση των επιτόπιων ελέγχων, που είναι απαραίτητη για την ε, ε, αποτελεσματική διαχείριση των ε, κινδύνων σε ό,τι αφορά την ε, αξιοπιστία, τη δήλωση αξιοπιστία, τη διαχειριστική δήλωση αξιοπιστία, θα πρέπει να ποσοτικοποιούνται οι δημοσιονομικέ συνέπειε και οι αδυναμίες του συστήματο να εντοπίζονται και με βάση την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου οι περισσότερες διορθώσεις είναι καταποκοπή διορθώσεις στη Γεωργία. Κάτι που αφισβητείται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και προτείνω να ευθυγραμμίσουμε αυτή την πολιτική με άλλα όργανα ε, μεικτής διαχείρισης ε, της συνοχής και να χρησιμοποιούμε στατιστικά ακριβή δείγματα σε μεγαλύτερο βαθμό, ώστε να περιορίσουμε τις καταποκοπή διορθώσεις και να έχουμε καλύτερη, πιο υγιή βάση για τις ε, αποφάσεις ε, της συμμόρφωσης. Ό,τι αφορά τα συστήματα ελέγχου και τις κυρώσεις, θέλω να αυξηθούν ε, τα ποσοστά μειώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επανειλημμένης μη συμμόρφωσης ή εσκεμμένης η εκπροθέσεως μη συμμόρφωσης, γιατί πιστεύω ότι τα μέτρα αυτά θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και θα συμβάλλουν στην καλύτερη καταπολέμηση, ιδιαίτερα της ε, εσκεμμένης μη συμμόρφωσης. Έχω κάποιες ερωτήσεις και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε πολύ επικοδομητικέ συζητήσει με του εκπροσώπου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα ήθελα και πάλι να σα ρωτήσω, με βάση τι ειδικέ εκθέσει του ε, ελεκτικού συνεδρίου 92% των διορθώσεων ε, είναι κατά αποκοπή διορθώσεις. Τι συγκεκριμένα μέτρα πιστεύω ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να, έχουμε, να χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο στατιστικά ακριβή δείγματα και σε ό,τι αφορά την εξαίρεση των μικρών γεωργών, των μικροκαλλιεργητών. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να εξαιρούνται από τη διαδικασία της πολλαπλής συμμόρφωσης. Στο σχέδιο γνωμοδότησης ε, τάσσομαι υπέρ των συστάσεων του Ελεκτικού Συνεδρίου για μη εξαίρεση των μικροϊών γεωργών και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι συγκεκριμένους μηχανισμούς μπορεί να προτείνει προκειμένου και αυτοί οι μικροκαλλιεργητές να υπόκεινται σε έλεγχο με κατάλληλες διαδικασίες. Και τελευταίο θέμα Γενικά, ο κανονισμός προβλέπει μείωση του αριθμού των ελέγχων σε μερικές περιπτώσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις. Πώς όμως μπορούμε να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικό έλεγχο και διασφάλιση της γενική ποιότητα του ελέγχου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σιγήτρια για την παρουσίαση των τροπολογιών σας. Και με ναι, έγκαιλε, θέλετε να λάβετε το λόγο εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την κυρία Ιβανόβα για την έκθεσή τη και για την καλή επαφή που είχαμε και την καρποφόρα συζήτηση για το σχέδιο γνωμοδότησης που έχετε προετοιμάσει. Μιλάμε για το επίπεδο δαπανών, όπω προτείνει η Κομισιόν, περίπου 60 δις ευρώ ετησίω προβλέπονται από τον που και αυτό ορίζεται στον οριζόντιο, στην πρόταση για τον οριζόντιο κανονισμό. Αυτό σημαίνει πω είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο και πραγματικά αξίζει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι όσο γίνεται καλύτερο. Η γνωμοδότηση είναι πολύτιμη ε, και περιλαμβάνει πολλά σημεία τα οποία, ε, με τα οποία συμφωνούμε. Τις τροπολογίες 4, 6 και 12 πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφέρω εδώ. Ε, μπορούμε επίσης να δούμε θετικά και άλλες τροπολογίες, αν και βλέπουμε και να υπάρχουν κάποια κενά όπως στις τροπολογίες 1, 7 και 11 και φυσικά είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τους δισταγμούς μας. Οι τροπολογίε όπου έχουμε πιο σοβαρού δισταγμού σχετίζονται καταρχήν με αυξημένη συμμετοχή τη Κομισιόν στη διαχείριση του CRP από τα κράτη-μέλη. Είναι οι 2, 3, 10 και οι 14. Ένα παράδειγμα που σχετίζεται με την τροπολογία 2. Αυτό που προτείνεται στο σχέδιο χρηματοδότηση είναι βασικά ότι η Κομισιόν δίνει μια εκ των προτέρων έγκριση τη διαδικασία διαπίστευση, στην οποία προβαίνουν τα κράτη-μέλη. Το βασικό επιχείρημα από θεσμική άποψη είναι ότι εδώ κινούμεθα σε ένα τομέα που ονομάζεται κοινή διαχείριση και που συμπεριλαμβάνεται στο δημοσιονομικό κανονισμό και σύμφωνα με αυτόν σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη διαχειρίζονται τα κονδύλια και η Κομισιόν έχει εποπτικό ρόλο, ιδιαίτερα ex post. Αυτή την αρχή λοιπόν θα την διαδράσαμε, θα την παραβιάζαμε αν η Κομισιόν άρχιζε να ασχολείται εκ των προτέρων. Πράγμα που σημαίνει ότι μετά θα βρισκόταν με δεμένα τα χέρια στους ε, εκ των υστέρων ελέγχους. Ε, δεν θέλουμε να ε, το κάνουμε αυτό. Να προσθέσω ότι έχουμε 81 γραφεία, γραφεία τοπικά, οργανισμούς πληρωμής δηλαδή ε, και αν γίνει μια τέτοια διαδικασία θα καθυστερούσε η διαδικασία και θα ε, περιορίζονταν οι δυνατότητες του προσωπικού. Θα ήθελα μάλιστα να σας παραπέμψω στο γεγονός ότι η Γενική Διεύθυνση για Regio εγκατέλειψε την ιδέα της προηγούμενης έγκρισης διότι είδα στην διαπίστωση ότι στην προηγούμενη διαδικασία καθυστέρησε αυτό το ξεκίνημα των προγραμμάτων. δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Όλοι μιλάνε για ανάπτυξη και θέλουμε όσο γίνεται να μπορέσουμε να εμβάσουμε αυτά τα χρήματα επί τη βάση των όσων έχουν σχεδιάσει τα κράτη-μέλη σε ε, συμφωνία βέβαια με τους ισχύοντες κανόνες. Αυτό δεν σημαίνει πως η Κομισιόν δεν εξετάζει τη διαδικασία διαπίστευσης διαρκώς ελέγχουμε τα σώματα διαπίστευσης στα κράτη-μέλη και βρίσκουμε κάποιες ανομαλίες όταν τις βρούμε αυτές ε, ζητάμε από τα κατημέρια να ελέγξουν, να θέσουν υπό διαδικασία ελέγχου τους οργανισμούς πληρωμής ή πιστοποίησης ε, ό,τι κάνουμε μέχρι σε εξπόστε σημαίνει φυσικά πως έχει αντίκτυπο και στο μέλλον. Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι για την επόμενη περίοδο δημοσιονομικής, ε, δημοσιονομικού προγραμματισμού δεν θα πρέπει να ξαναγίνουν όλες οι πιστοποιήσεις. Τα οι περισσότεροι οργανισμοί θα παραμένουν ως έχουν, απλώς θα πρέπει να προσαρμοστεί η πιστοποίηση στα νέα μέτρα και στις νέες διατάξεις χρειάζεται σαφής διαχωρισμός ευθυνών ανάμεσα στη διαχείριση των κρατών μελών και τον έλεγχο της ε, Κομισιόν. Κάποια άλλα στοιχεία τώρα. Τροπολογία υπαριθμών 5. Εδώ ίσως υπάρχει κάποια, κάποια ε, παρεξήγηση. το θέμα των οργανισμών πληρωμών δεν έχει σχέση με τους οργανισμούς πληρωμής ε, στον δημόσιο τομέα. Απλώς υπάρχει κάποια παρεξήγηση και πρέπει να διευκρινιστεί η κατάσταση. Η ε, τροπολογία 8 αφορά τον υπολογισμό των δημοσιονομικών διορθώσεων. Ε, ε, συμφωνώ μαζί σου ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε όσο γίνεται από συνολικές διορθώσεις που πολλές φορές σημαίνει πως είναι ποινές. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες για να το επιτύχουμε αυτό. Και τώρα, στο πλαίσιο του οριζόντιου ε, κανονισμού, θέλουμε να φτιάξουμε μια νέα διαδικασία μαζί με τους οργανισμούς πιστοποίησης που θα μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε πιστοποιημένα ποσοστά σφάλματα, σφάλματος που θα είναι πιστοποιημένα από τα συγκεκριμένα αρμόδια όργανα ε, αρμόδια, για, για αυτούς τους σκοπούς είναι ο ρόλος της Κομισιόν να ε, προβαίνει σε στατιστικό δείγμα, δειγματοληψία και πάλι εδώ δεν είμαστε εμείς που το κάνουμε αυτό, τα κράτη-μέλη είναι που κάνουν δειγματοληψία. Η Κομισιόν φτιάχνει τους κανόνες για την επιλογή του δείγματος και αυτό κάνουμε. Ακολουθούμε ένα πολύ λεπτομερές έγγραφο εργασίας το οποίο θα ολοκληρωθεί μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές και θα σταλεί στο Ευρωκοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη ώστε να δείτε καλύτερα ποια είναι, ποια είναι τα προγράμματα της Κομισιόν, τα σχέδια μάλλον της Κομισιόν. Τροπολογία 9 νομίζουμε ότι είναι σε αντίφαση με την 8, γιατί οι καταποκοπήν διορθώσεις δεν μπορούν να αντικατασταθούν από υπολογισμένε διορθώσεις μόνο επί τη βάση ε, τεκμηρίωσης από το κράτη-μέλη. Ε, δεν θα ήταν αρκετό κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γίνουν επιτόπου έλεγχοι. Τροπολογία 14 και 17 και 18 που αφορούν, αφορούν όλες την πολλαπλή συμμόρφωση. Κυρία Ιβάνοβα, αναφερθήκατε στην πρόθεσή σας ή στην επιθυμία σας να ενισχυθούν οι ποινές σε αυτούς τους τομείς, οι κυρώσεις. Εδώ μιλάμε για κυρώσεις στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης. Όσον αφορά την τροπολογία 14, προτείνεται η Κομισιόν να δώσει μια εξασφάλιση πως ορισμένες περιφέρειες με μικρούς ε, γεωργούς δεν θα αποκλείονται σε μεγάλο βαθμό από την πολλαπλή από το σχέδιο πολλαπλής συμμόρφωσης. Η τροπολογία όπως έχει συνταχθεί είναι πολύ δύσκολο να δυσχεραίνει μάλλον τη λειτουργία της Κομισιόν. Πώς μπορούμε να δώσουμε τέτοια εξασφάλιση όταν ταυτόχρονα ο νομοθέτης έχει φτιάξει ένα κανόνα που λέει ότι σύμφωνα με το σχέδιο για τους μικρούς ε, γεωργούς ε, η πολλαπλή συμμόρφωση δεν ισχύει. Τότε βέβαια η Κομισιόν δεν θα αρκούσε. Δεν θα μπορούσε μάλλον να συμμορφωθεί προς ένα τέτοιο κανόνα. Και όσον αφορά την εξαίρεση των μικρών γεωργών από την πολλαπλή συμμόρφωση, να αναφέρω Μόνο μία παρατήρηση έχω να κάνω ακόμα. Τροπολογίες 17 και 18. Εδώ προτείνεται ορισμένες κυρώσεις να είναι τουλάχιστον 5%. Αυτό σημαίνει πως ποινές κάτω από αυτό το ποσοστό δεν θα μπορέσουν να εφαρμοστούν ακόμα και σε περιπτώσεις μικρότερων παραβιάσεων ή μικρότερης θα έπρεπε να εφαρμόσουμε πολύ δυσανάλογες κατά τη γνώμη μας ποινές. Και εδώ θα πρέπει μαζί λίγο να δούμε τι διατάξεις αυτές για να ε, συμμορφωθούν προς την αρχή της αναλογικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. κύριε Ρούντοφ Μέγκελε για τη συμβολή σας. Πριν να δώσω το λόγο στην συγκήτρια, θα καλωσορίσω μια αντιπροσωπεία από την Ουγκάντα, αν ε, μου είπαν σωστά. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού και τώρα θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, Ηλιάνα Ιβάνοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μέγκελε για τις παρατηρήσεις τους. Clarify any issues that need to be clarified. Όντως διευκρινίστηκαν ε, ορισμένα σημεία που είχαν ε, μείνει εκρεμή. Έχω και εγώ μερικά σχόλια με το δικό σα. Σε ό,τι αφορά την ευθύνη, νομίζω ότι ο ίδιος δημοσιονομικός κανονισμός προβλέπει ότι σε έσχατο βαθμό αρμόδια για την ε, εκτέλεση του προπολογισμού είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή έχει και τον τελικό λόγο σε ό,τι αφορά την εκτέλεση. Γι' αυτό και ζητούμε κάτι παραπάνω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο ευθυγραμμίζεται με το δημοσιονομικό κανονισμό. Σε ό,τι αφορά την εξάντε έγκριση, την εκ των προτέρων έγκριση, γιατί να μην μπορούμε να εφαρμόζουμε και τέτοιο εκ των προτέρων έλεγχο. Κάτι τέτοιο ήδη ίσχυσε για κάποιους οργανισμούς πληρωμής και τη διαπίστευσή τους, για τα προενταξιακά κονδύλια. Και μάλιστα η τροπολογία, έτσι όπως έχει διατυπωθεί, δεν ζητά έλεγχο όλων των οργανισμών πληρωμής, αλλά με βάση τον κίνδυνο και το ποσοστό κινδύνου είναι πολύ μικρό τελικά ο αριθμό των οργανισμών πληρωμή που θα πρέπει να ελεγχθούν με αυτόν τον τρόπο που ζητούμε, εκ των προτέρων δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά έγκυρα δείγματα, με εκπλήσει το γεγονό ότι θεωρείται ανέφικτη αυτή την πρόταση. Γιατί όμως γίνεται κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο στο Ταμείο Συνοχή, ενώ για το Γεωργικό Ταμείο θεωρείται ότι είναι ανέφικτο. Δεν καταλαβαίνω τη διαφορά. Παρακαλώ, θα ήθελα και εδώ κάποιες εξηγήσει. Πάντω σα ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε έτσι τελευταία στιγμή ε, και θα σταματήσω εδώ τα σχόλιά μου. Ευχαριστώ τη τη της γνωμοδοτήσεω, κυρία Ιβάνοβα. Ρωτώ και πάλι τον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου αν επιθυμεί να τοποθετηθεί. Όχι, πολύ καλά. Και τότε εδώ έληξε και αυτή η συζήτηση. Προβλέπεται προθεσμία καταθέσεις τροπολογιών μέχρι την 17 η και ψηφοφορία επί του κειμένου στις 17 Ενάτου. Έχουμε εξαντλήσει και την ημερήσια διάταξή μας. Ευχαριστώ όλες και όλους, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες της Γραμματείας, τους εκπροσώπους ε, της Κομισιόν, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και των άλλων ενδεχομένως ε, οργάνων διευθύνσεων που έλαβαν μέρος στην ε, συνεδρία. Ευχαριστώ.